Uh, dear colleagues, dear friends. Κυρίες και κύριοι, έχουμε βεβαίως την ημερήσια διάταξή μας. Θα χαρώ πολύ να την εγκρίνετε, αλλά να πω πρώτα, ή μάλλον να ζητήσω συγγνώμη πρώτα για την καθυστέρηση, όμως ε, διεξήχθησαν πολλές συζητήσεις στην συνάντηση των συντονιστών μας και ελπίζω να μπορέσει να ολοκληρωθεί η συνάντησή μας μέχρι τις 12.30. Όμως τώρα στην αρχή έχω ένα θλιβερό νέο διότι με μεγάλη θλίψη σας πληροφορώ ότι ο συνάδελφός μας και αντιπρόεδρος μας Μύροσλαβ Ράνσντορφ απεβίωσε δυστυχώς στις 22 Ιανουαρίου. Από τότε που πρωτεκλέχθηκε Ευρωβουλευτής το 2004 πολλοί, πολλοί από εμά τον θυμόμαστε πολύ καλά ο Μύροσλαβ υπήρξε ενεργό μέλος της Επιτροπής ΙΤΡΕ συνεχώς και τα 12 αυτά χρόνια. Το έργο του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμανε μια μακρά πολιτική σταδιοδρομία στην διάρκεια της οποίας ήταν και για 8 χρόνια βουλευτής στην Τσεχική Βουλή μεταξύ 1996 και 2004 δύο ε, συνεχείς θητείες και πριν από αυτό στην Τσεχοσλοβακική Ομοσπονδιακή Συνέλευση το 1992 για δύο χρόνια δύο πολύ σημαντικά χρόνια για την ε, Τσεχοσλοβακική Ομοσπονδιακή Συνέλευση. Ο Λαβ ήταν πραγματικός πολιτικός, πάντοτε αποφασισμένος να εξηγήσει και να υποστηρίξει τις ιδέες του. Θα τον θυμόμαστε πάντα σαν έναν άνθρωπο γεμάτο θέρμη και καλό συνάδελφο. Είμαι βέβαιος ότι μοιράζεστε τα ίδια συναισθήματα μαζί μου. Για πολλά χρόνια τον βασάνιζε η ασθένεια. Από την αρχή που εξελέγει Ευρωβουλευτής, το ένιωθε και κανείς. Ήταν και αντιπρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ενέργειας και μάλιστα πολύ δραστήριος και παρόν στις συναντήσεις μας στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες και στην προηγούμενη θητεία, αλλά σε τούτην εδώ τη θητεία μάλιστα ήταν και αντιπρόεδρος και ιδιαίτερα δραστήριος. Ο Μυροσλάβ ε, αφήνει πίσω την σύζυγο και τη θηγατέρα του, προς τις οποίες εκφράζω τα ειλικρινέστατα συλληπιτήριά μας. Υπάρχει και βιβλίο συλληπιτηρίων στην ε, μνήμη του Μύροσλαβ Ράνστορφ. Είναι ανοιχτό στο επίπεδο αυτό εδώ στο κτίριο του Κοινοβουλίου, λίγα μέτρα πιο έξω από την αίθουσά μας και θα είναι και έξω από την αίθουσα του ημικυκλίου στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα. Άρα και εδώ στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, προτείνω ενός λεπτού σιγή. Εις μνήμην του φίλου μας. Thank Σας ευχαριστώ. Είναι η υποχρέωσή μου τώρα να μεταβώ στην ε, διάσκεψη των Προέδρων. Θα χρειαστεί λοιπόν να εγκαταλείψω την συνεδρίασή μας. Θα είμαι όμως και πάλι εδώ στις 3, στο δεύτερο μέρος της ε, συνάντησής μας. Έτσι είναι στις 3. Θα παραδώσω τα ενία της συζητήσεως στον αντιπρόεδρό μας, κύριο Headcamp. Okay, let's uh, Ας συνεχίσουμε. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή της οδηγίας για την αποδοτικότητα της ενέργειας και χωρίς περισσότερα λόγια να προτείνω να αρχίσει ο κύριος Μάρκους Πίπερ του Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ, αγαπητέ Πρόεδρε. Ελπίζω το μικρόφωνο μου να λειτουργεί. Έχουμε όντως στα χέρια μας ένα νέο εργαλείο ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή την έκθεση εφαρμογής, όπου μπορούμε εμείς να σημειώσουμε τις απόψεις μας αν όντω έχει αποδώσει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αν σημειώνονται προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή αυτή και αν από τη δική μας σκοπιά υπάρχουν ιδέες που θέλουμε να υποβάλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για την επανεξέταση της οδηγίας η οποία επίκειται το φθινόπωρο. Επ' αυτού μπορώ να σας πω ότι βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από την έναρξη της ε, παρούσας κοινοβουλευτικής περίοδου, διότι μπορούμε να διεξαγάγουμε δικές μας μελέτες και έρευνες και αυτό το έχουμε ήδη πράξει σε μεγάλο βαθμό για τούτο εδώ το θέμα, την αποδοτικότητα της ενέργειας. Ευχαριστώ και τους και με τους οποίους ήδη έχω συναντηθεί και ευχαριστώ πολύ και τους διάφορους ενδιαφερομένους. Μάλιστα διεξήχθηκε ειδική ακρόαση. Υπάρχει λοιπόν έντονο ενδιαφέρον. Τώρα επί του ουσιώδους περιεχομένου. Πρώτα, μια προκαταστική παρατήρηση. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά τους στόχους της προστασίας του περιβάλλοντος, έχουμε εξέχουσα θέση. Από το 1990 έχουμε μειώσει τις εκπομπές των διαφόρων οξυδίων του άνθρακα κατά 23%. Ταυτόχρονα το ΑΕΠ της Ευρώπης αυξήθηκε κατά 46%. 22% κάτω το διοξείδιο του άνθρακα, 46% πάνω το ε, ε, εθνικό προϊόν. Πάνε καλά τα πράγματα λοιπόν. Ναι, μεν πάνε καλά τα πράγματα, αλλά ποιο είναι το τίμημα της ανταγωνιστικότητας και ποια είναι η γραφειοκρατία που έχει αναπτυχθεί. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτή την θετική πορεία για το περιβάλλον, θα χρειαστεί κάποια πράγματα να αλλάξουμε. Και <clears throat> ιδίω την αλληλοεπίδραση των υφιστάμενων νομοθετημάτων που καμιά φορά μάλιστα είναι και αντιφατικά. Έχω λοιπόν πολλές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα θέσω πρώτα ορισμένες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ε, ε εφόσον γίνει υποχρεωτική η εξοικονόμηση ενέργειας για τους παρόχους ενέργειας. Αυτό δεν έχει ε, συνέπειες και στο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Δεύτερο, εάν υπάρξει υποχρεωτική εξοικονόμηση πάλι, τότε η επέκταση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν παρεμποδίζεται. Υπάρχουν πάροχοι Ενέργειες οι οποίοι έχουν ειδικευτεί σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θέλουμε λοιπόν να του επιβάλλουμε πράγματι και σε αυτούς ε, ε, υποχρεωτικά την εξοικονόμηση ενέργειας. Τώρα, eco-design και ε, διάφορες ετικέτε, επισημάνσει για την ενέργεια στα κτίρια κτλ. Δεν έχουν επίσης και αυτά τις ίδιες επιπτώσεις, δηλαδή μήπως κάνουμε επικάλυψη προσπαθειών. Τρει και τέσσερι φορέ Έχουμε δηλαδή και την οδηγία ED4 που έχει του ίδιου στόχου. Ήδη ισχύει από το 2014 η οδηγία για την αποδοτικότητα τη ενέργεια, Οι περισσότερε από τι χώρε μέλη αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην εφαρμογή τη και αυτό το επικρίνουμε. Και με την παλαιότερη οδηγία περί σε πέντε χώρε μέλη και σημαντικέ μάλιστα αντιμετωπίζονται σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή τη. Ακολουθεί τώρα η επόμενη ερώτησή μου. Γιατί Παρ' όλα αυτά πετυχαίνουμε τους στόχους της εξοικονόμησης ενέργειας. Βρισκόμαστε σχεδόν, δηλαδή προχωρούμε προς το 100% παρόλο που δεν αποδίδουν οι οδηγίες. Μήπω υποτιμούμε την ε, επίπτωση άλλων νομοθετημάτων. Μήπως υποτιμούμε και το ίδιο συμφέρον των καταναλωτών οι οποίοι επενδύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και χωρίς υποχρεωτικά μέτρα. Έρχομαι τώρα στην ουσία, στον πυρήνα έχουμε 2.000 υποχρεωτικές αναφορές για κρατικές αρχές κλπ που σημαίνουν μια τεράστια γραφειοκρατία. Κάπου έχουμε ξεπεράσει κάποιες κόκκινες γραμμές. Και έρχεται τώρα και η κυκλική οικονομία με νέες ποσοστώσεις για ε, πρώτες ύλες, για ενέργεια κτλ. Έχω και εδώ κάποια νούμερα. Από το 2002 η χρήση πρώτων υλών στην Ευρώπη, η χρήση πρώτων υλών, έχει μειωθεί κατά 30% ανά, ανά μονάδα του ΑΕΠ. Ανά μονάδα του ΑΕΠ λιγότερο 30% χρήση πρώτων υλών. Και αυτό είναι καλή είδηση. Νομίζω ότι αυτή τη θετική πορεία για το περιβάλλον πρέπει να τη συνεχίσουμε. Χωρίς όμως να επιβαρύνουμε υπερβολικά τις καλές προθέσεις με γραφειοκρατία. Έχουμε εθνικά σχέδια, οδικούς χάρτες για την εξυγένση των κτηρίων, για την ε, βελτίωση των λογαριασμών, έχουμε τους ελέγχους ενέργειας, audit δηλαδή, την διασύνδεση ε, της παραγωγής ενέργειας με τη θέρμανση κλπ. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Και βεβαίως όντως δεν έχει αρχίσει να αποδίδει ακόμα η εφαρμογή της οδηγίας. Όμως θέτω και πάλι την ερώτηση. Αυτές οι καταρχήν θετικές ιδέες Μήπως μπορούν να επιτευχθούν και με λιγότερη γραφειοκρατία και με λιγότερους ελέγχους. Μήπως μπορούν να ενταχθούν καλύτερα σε άλλες υφιστάμενες οδηγίες ε, οι νομοθετικές αυτές προβλέψεις. Μήπως μπορεί να ολοκληρωθεί και να συμπληρωθεί το ε, ETS, το σύστημα εμπορίας. <clears throat> Ακόμη και το χαρακτηριστικό, το σήμα CE δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτό και να συμπληρωθεί με <clears throat> μια σφραγίδα η οποία θα μπαίνει πάνω σε όλα τα προϊόντα που εξοικονομούν ενέργεια κτλ. Κάτι το οποίο μας, θα μας εξυπηρετήσει. Νομίζω ότι κάπου έχουμε χαθεί μέσα σε αυτή την εφορία που μας διακατέχει λόγω των ποσοστώσεων κλπ. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιβαρύνουμε περισσότερους καταναλωτές και τους παρόχους. Με μεγάλη μου χαρά λοιπόν θα ε, συνεχίσω την συζήτηση αυτή μαζί σας τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, αλλά και την συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα, αλλά στηρίσουμε και το όριο ε, του χρόνου αγορεύσεως, λέει ο πρόεδρο. Πρόεδρος. Εσείς τα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Χόντσον, έχετε 10 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και είναι μια καλή χρονική στιγμή και χαιρετίζουμε το γεγονό ότι το Κοινοβούλιο αξιολογεί το ζήτημα από ό,τι κατάλαβα θα, είχε, θα ψηφίσετε στις 24 Μαΐου. Ακριβώς αυτό το τμήμα της ε, νομοθεσίας επανεξετάζομαι με μια προσπάθεια να επανέλθουμε με πρόταση το Σεπτέμβριο. Επομένως το χρονοδιάγραμμα λειτουργεί. Η οδηγία ενεργειακής απόδοσης είναι το ευρύτερο, το γενικότερο πλαίσιο για τη δουλειά μας. Το υιοθετήσαμε διότι εκείνη τη στιγμή οι προβλέψεις ήταν ότι θα επιτυγχάναμε μόνο το τους 10 από τους 20 ποσοστίες μονάδες που είχαν θέσει ως στόχο και εμείς βρισκόμαστε εν μέσω της αξιολόγησης της οδηγίας δεν μπορώ να τοποθετηθώ τελεσίδικα για τη διαδικασία αυτή όπως και εσείς δεν μπορείτε αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είχαμε υποβάλει έκθεση προόδου το περασμένο φθινόπωρο όπου συνολικά δείχνει ότι η πρόοδος στην ενιακή απόδοση είναι πολύ καλή. Τα κράτη-μέλη δίνουν ενδείξεις για 19 με 20%. Αυτό βεβαίω επί τη βάση των όσων γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή για την υλοποίηση στα κράτη-μέλη. 18 με 19% και από, και ό,τι μας λέει η ανάλυση μας θα επιτύχουμε τελικώς το 20% εάν υλοποιήσουν πλήρως το νομοθετικό πλαίσιο που έχουμε αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη δυσκολεύονται όχι επειδή ε, κάτι τέτοιο είναι μια επακθής ευρωπαϊκή υποχρέωση, κατά την άποψή μας, και όχι επειδή είναι πράγματα που δεν θέλουν να κάνουν, θέλουν να τα κάνουν. Ο λόγος που δυσκολεύονται είναι ότι ο στόχος είναι δύσκολος. Η εκεί απόδοση είναι δύσκολος στόχος. Και είναι κάτι που πρέπει να προχωρήσει κανείς κτίριο-κτίριο. Δεν υπάρχει κάποια λύση που να μας επιτρέπει να προχωρήσουμε ομαδικά όπως να πούμε ότι θα θέσουμε την τάδε υποχρέωση στον τάδε τομέα. Έχει όμως γίνει πρόοδος, η οποία πρόοδος έχει επιτευχθεί μετά από σκληρές προσπάθειες και αυτό δείχνει τη βούληση των κρατών μελών. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε την μεταγραφή, την μεταφορά και η εικόνα είναι ότι πολύ σπάνια μεταγράφονται όλα τα στοιχεία των νομοθετημάτων απολύτως εγκαίρως, αλλά με τις διαδικασίες παραβίασης που υπάρχουν, κάθε στοιχείο της οδηγίας που ε, ήταν να μεταγραφεί και να, να εφαρμοστεί, έχει εφαρμοστεί τελικώς. Μέχρι τις 30 Απριλίου του 2013 ήταν η προθεσμία για τους στόχους απόδοσης και εντος 2 2-3 μηνών το είχαν πράξει ακόμα και οι πιο καθυστερημένοι. Για τους υπόλοιπους στόχους εντός 5 μηνών από την προθεσμία από το τέλος του ιδίου έτους ήταν ο επόμενος στόχος δηλαδή. Εν πάση δηλαδή, ακόμα και με κάποιες καθυστερήσεις όλοι κρατάνε τους στόχους της οδηγίας. Και αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε την ε, δουλειά μας για την ε, μεταφορά και για στοχευμένα στοιχεία, πτυχές της οδηγίας. Δεν έχω δηλαδή μια απόλυτη εικόνα για τη συνολική πρόοδο της οδηγίας. Βεβαίως και παρακολουθούμε το στόχο, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Οκτωβρίου του 2014, και για ένα συνολικό στόχο 40% υλικό, όπου πρέπει να αναθεωρήσουμε τις διατάξεις των άρθρων της οδηγίας για να δούμε τα άρθρα δηλαδή 1 και 3, το άρθρο 6 για τις δημόσιες προμήθειες, το άρθρο 7 για τις υποχρεώσεις νεακή απόδοσης και εναλλακτικέ. Και εξετάζουμε και δύο δέσμες άρθρων, 9-12 για την ε, επιμέτρηση και το 15, 8 για ζήτηση και προσφορά σχετικά με το όσο γίνονται στα πλαίσια της πρωτοβουλίας νεαϊκού σχεδιασμού. Τις υπόλοιπες διατάξεις δεν τις επανεξετάζουμε. Είχαμε κάνει μια, αυτή τη στιγμή μάλλον όπως σας έλεγα κάνουμε, τρέχουμε μια αξιολόγηση. Ελπίζω ότι αυτή θα δημοσιευθεί μαζί με τις ε, ε, ε συνυπικουρούσες εκθέσεις το Μάρτιο και αυτό ελπίζουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι ένα σημαντικός πολύτιμος πόρος για όλους εσάς. Μπορώ να σας δώσω κάποια προκαταρτικά στοιχεία των μελετών αυτών γιατί εξεκολουθεί η δουλειά αυτή. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 6 δημόσιες προμήθειες, η ενδείξη είναι ότι είναι υπερβολικά νωρί για να σκεφτούμε να τροποποιήσουμε το πλαίσιο γιατί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για ένα αποτελεσματικό κεντρικό κυβερνητικό καθεστώς δημοσίων προμηθειών στα κράτη-μέλη. Στο άρθρο 7 η πρώτη ένδειξη είναι ότι αυτό το άρθρο, ότι μάλλον τα σχέδια που έχουν τα κράτη-μέλη, εφόσον λειτουργήσουν, θα οδηγήσουν στους στόχους ενεργειακής απόδοσης, ε, αποταμίευσης στην ουσία, σχετικά με τις εναλλακτικές ε, πηγές που έχουμε θέσει ως στόχο. Δευτερευόντως, 16 κράτη-μέλη χρησιμοποιούν τις υποχρεώσεις συνεργικής απόδοσης για μέρος της εφαρμογής τουλάχιστον, τα υπόλοιπα 12 μόνο εναλλακτικές λύσεις και τα υπόλοιπα μεικτή προσέγγιση. In particular, have a relatively low... Όλα αυτά έχουν σχετικά χαμηλό διοικητικό κόστος, σύμφωνα με το δεδομένο που έχουμε. Δηλαδή, για τέσσερα κάτι μέλη έχουν κρατήσει το κόστος κάτω του 0, 2, 3 ή 4 του συνολικού του προγράμματος. Και για ένα κράτος μέλος λίγο άνω του 1% του συνολικού κόστους. Σχετικά με ανταλλάξιμες υποχρεώσεις. Για τις εναλλακτικές ε, προσεγγίσεις δεν έχουμε το διοικητικό κόστος και για το κόστος για τους πολίτες εφόσον τεθεί μια υποχρέωση επί συγκεκριμένου προϊόντος, συγκεκριμένης ε, ενιακής πηγής αντισταθμίζονται τα ωφέλη για τους πολίτες με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν. Και το τελικό αποτέλεσμα, ο τελικός ολογισμός είναι τελικά θετικός για τους καταναλωτές. Εκεί κάπου βρισκόμαστε στην ε, αναθεώρηση του 7 Έχουμε θέματα συμπληρωματικότητας, διπλής καταμέτρησης. Πρέπει να δούμε κάποια τέτοια θέματα για να απλουστεύσουμε τι διατάξει περαιτέρω για να είναι σαφείς και αποτελεσματικές. Αλλά και με την παρελούσα μορφή τους η μελέτη λέει ότι λειτουργούν συνολικά καλά. Για τη δημόσια διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί αύριο, 29 Ιανουαρίου, το 71% των απαντήσεων βρίσκουν το άρθρο 7 αποτελεσματικό, το 73% θεωρεί ότι πρέπει να επεκταθεί πέραν του 2020 και οι περισσότεροι εξεργούν θετικά τις περισσότερες στοιχές. <clears throat> Υπάρχει ευρία στήριξη. Βεβαίως το να μετράμε αριθμό στη δημόσια διαβούλευση δεν είναι αναγκαστικά η καλύτερη λύση. Για τις επικαλύψεις ή μάλλον για το κοινό συμφέρον με την ε, κοινή αγορά ενέργειας. Ε, ε, συνεχίζουν οι μελέτες, δεν έχω προκαταρκτικά συμπεράσματα εδώ. Απλώς να βεβαιώσω όλους ότι για τα άρθρα 1 3 ε, δεν εξετάζουμε μόνο το, τη δέσμη στο 27-30% αλλά και τις υπόλοιπες δέσμες. Τώρα, για τις ελάχιστες προϋποθέσεις αγοράς νέων προϊόντων και ετικετοθεσία σχετικά με την ενιακή της απόδοση. Το ίδιο κάνει η νομοθεσία ε, των ε, κτηρίων με ελάχιστες προϋποθέσεις της ανακαίνησης κτλ. Αυτό που κάνει η οδηγία ενιακής απόδοση σε όλους τους τομείς είναι ότι αυξάνουν το ποσοστό στο οποίο προχωρούμε σε νέες ανακαινήσεις, το ποσοστό στο οποίο προχωρούμε σε αγορά νέων προϊόντων με νέα επισήμανση. και την ερώτηση του πώς επιτυχάνουμε τους στόχους μας με τις δυσκολίες εφαρμογής, η εκτίμησή μας για το 18-19% αποτέλεσμα βασίζεται στο ρυθμό στον οποίο αυτή τη στιγμή εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη την οδηγία. Και νέα με καθυστερήσεις, δυστυχώς, αλλά την εφαρμόζουν. Περιμένουμε ενδιαφέρον την δική συζήτηση. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπενθυμίζω ότι στην διάρκεια των συναντήσεων Ήτρε στις 16 και 17 Μαρτίου θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε την έκθεση αυτή. Για την ώρα προτιμώ να εστιάσουμε, να εστιάσουμε στις πολλές ερωτήσεις που έχουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα παρακαλέσω τώρα τον κύριο Πόχε των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ήταν σημαντική ευφυής και στρατηγική απόφαση για την απόδοση, για την ενεργειακή απόδοση και έχει οδηγήσει και σε εξοικονομήσεις και μπορεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, να ενισχύσει την ασφάλεια των προμηθειών αφού θα χρειάζονται λιγότερο πετρέλαιο και άλλες ενέργειες, μειώνει το κόστος για τα νοικοκυριά, σημαντικό αυτό για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματο και τέλος είναι και από τους πιο φθηνούς τρόπους για να μειωθούν οι εκπομπές ιδιοξιδίου του άνθρακο. Βεβαίως είναι κρίμα που δεν πρόκειται να επιτύχουμε όλους τους στόχους της ενεργειακής απόδοσης μέχρι το 2020 αν και έχουν γίνει σημαντικές πρόοδοι. Έχουν γίνει όχι αμελητές μειώσεις της ενέργειας όπως δείχνει και η έκθεση πρόοδου της Κομισιόν. Και στην οικοδομή και στη βιομηχανία οι χώρες μέλη έχουν επιβάλει νέα μέτρα για την μείωση της ε, κατανάλωσης ενέργειας. Όμως αυτά δεν είναι επαρκή. Πάμε να φτάσουμε μόνο στο 18 με 19% για την ώρα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτό που χρειάζεται είναι να βάλουμε ξεχωριστούς εθνικούς στόχους. Η οδηγία προβλέπει έναν αριθμό μέτρων για να ενισχυθεί η μείωση της χρήσης ενέργειας. Αυτά όμως πρέπει να συνδυαστούν και με, άλλα, και με άλλους μηχανισμούς, δημοσιονομικούς και άλλους. Και τότε δημιουργείται ένα ευρύτερο πλαίσιο. Οι ελλείψεις που βλέπουμε τώρα οφείλονται στην έλλειψη εφαρμογίας της οδηγίας και στους όχι φιλόδοξους στόχους από την αρχή. Χρειάζεται να λάβουμε υπόψη και τις διάφορες περιστάσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες μέλη. Ταυτόχρονα η μεγάλη ευκαμψία που επιτρέπει η οδηγία είναι και η μεγάλη της αδυναμία. Έχω τώρα ορισμένα σημαντικά πράγματα. Πρώτον, θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα για να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των κτίριων. Το άρθρο 4 της οδηγίας απαιτεί από τις χώρες μέλη να καταγράψουν τα κτίρια τους και να προβλέψουν νέες στρατηγικέ για την ανακαίνισή τους. Ωστόσο υπάρχουν περιθώρια για μεγάλες βελτιώσεις γιατί ε, αυτό ο, ο τομέας φτάνει και στο 40% σε όλη την Ευρώπη. Το δεύτερο είναι η ευκαμψία, ιδίως για προγράμματα τα οποία ε, πρέπει να μπορούν να φτάσουν και μέχρι το 35% των στόχων. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί η ενεργειακή φτώχεια, θα επιτρέψει τα νοικοκυριά να βελτιώσουν την ενεργειακή τους ε, απόδοση και των κατοικιών τους και των άλλων κτηρίων επίση. Ο πρόεδρο διακόπτη, έχετε ξεπεράσει το χρόνο σας. Το 20% που βάζει ως στόχο η οδηγία ήταν σημαντικό πράγματι. Χρειάζεται όμως να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες που έχουν οδηγήσει στη μείωση της, ε, της ε, ενέργειας. Η θέσπιση διακόπτη πάλι ο πρόεδρος. Λυπούμε πολύ. Σκιώδης ηγητής είμαι κύριε πρόεδρε. Τώρα, η ομάδα Ευρωπαίων συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Δεν έχουμε εδώ τον σκιώδη ηγητή τους. Κύριε Πέτερσεν τώρα των φιλελευθέρων. Σας ευχαριστώ. Πράγματι βλέπω πολλές θετικές πτυχές της ε, ενεργειακής απόδοσης, όπως είπε και ο κύριος Πόχε, με την αύξηση της ε, ενεργειακής απόδοσης μειώνουμε τις εισαγωγές από Ρωσία και Μέση Ανατολή και μειώνουμε και τις ε, εκπομπές καυσαερίων. Πώς μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο, πώς μπορούμε να θεσπίσουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο να δίνει και κίνητρα για καινοτομία και να εξασφαλίζει την βέλτιστη δυνατή χρήση της ενέργειας. Πού θα βάλουμε προτεραιότητες, πώς θα χρηματοδοτήσουμε τις αναγκαίες επενδύσεις με χαρά μου βλέπω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τους σχετικούς υπολογισμούς που δηλαδή μπορούν να επέλθουν βελτιώσεις. Και χαίρομαι που τα βλέπει αυτά σε ευρύτερο πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε μια συνολικότερη νομοθεσία που μπορεί να επιτρέψει να επιτεθούν οι στόχοι που ανέφερα. Είναι δύσκολο το στάδιο αυτό να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά επιτρέψτε μου να σας αναπτύξω ορισμένες από τις δικές μας προτεραιότητες. Οι οικοδομές είναι πολύ σημαντικές διότι η θέρμανση ή ψήξη των κτηρίων καταναλώνει τεράστιο ποσοστό της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται στην Ευρώπη. Επομένω, σαφέστατα ο στόχος ανακαίνησης των δημόσιων κτηρίων είναι σημαντικός. Τα άθρα 4, 5 και 6 θα μας αναγκάσουν να διεξαγάγουμε πολύ ενδιαφέρουσε συζητήσει για το θέμα αυτό. Πρέπει επίσης να δούμε πώς θερμαίνονται ή ψύχονται τα κτίρια. Υπάρχουν πολλοί αποδοτικές λύσεις και, συνεχώ, και συνεχής καινοτομία στην αγορά. Όμως αυτά χρειάζονται πολύ συχνά σημαντικές επενδύσεις. Πώς θα τονώσουμε αυτές τις επενδύσεις, να μην λησμονούμε ότι εδώ τα πράγματα δεν είναι πράσινα μαύρα, πράσινα μαύρα ξαναλέω. Ορισμένοι είπαν ότι η ενεργειακή απόδοση μπορεί να εμφανιστεί και πολύ γραφειοκρατική. Όμως, εάν γίνει καλά, η πολιτική ενεργειακής απόδοσης μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και ταυτόχρονα να μας επιτρέψει να πετύχουμε τους περιβαλλοντικούς μας στόχους. Ελπίζω με τη συζήτησή μας να μπορέσουμε να διαλύσουμε κάποιους μύθους που σηκώνουν την άσχημη κεφαλή τους και από εδώ και από εκεί και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος και να προχωρήσουμε ίσως σε μια καλή συνεργασία με τους συνάδελφους. Ευχαριστώ. Γιάβορ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για, την, ε, για τις απόψεις της καθώς και τον κύριο Πίπερ. Σύντομες παρατηρήσεις. Ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού. Αυτά που αποφασίσαμε στο Παρίσι λένε ότι πρέπει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες μας, τις προσπάθειές μας για μείωση των εκπομπών καυσαερίων και όχι να τις επιβραδύνουμε. Η ενεργειακή απόδοση, όπως λέχθηκε, είναι από τις πιο χρήσιμες επιλογές για να μειώσουμε και τις ε, εκπομπές καυσαερίων, διοξείδιο του άνθρακος κυρίως. Αυτό όμως δεν είναι μόνο κατηγορική επιταγή για το περιβάλλον. Πιστεύω ότι η ενεργειακή απόδοση θα βοηθήσει την Ευρώπη σε πολλά και σε γεωπολιτικά, όπως είπε και ο κ. Πέτρασεν, η ενεργειακή απόδοση αυξάνει και την ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε πετρελαϊκά και άλλα σοκ. Νομίζω επίσης ότι η ενεργειακή απόδοση μπορεί να βελτιώσει και στην ανταγωνιστικότητα της, ε, των ευρωπαϊκών οικονομιών που ανησυχούν τον κύριο Πίπερ αυτά τα πράγματα, το άκουσα από τα όσα είπε. Πρέπει να οικοδομήσουμε μια ανταγωνιστική οικονομία στην Ευρώπη. Όμως η ενεργειακή αποδοτικότητα δεν είναι εμπόδιο. Είναι αντίθετα ένα εργαλείο που επιτρέπει την δημιουργία ε, ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Κάθε ευρώ που δαπανάμε εδώ στην ενεργειακή απόδοση μας εξοικονομεί 3 ευρώ από το κόστος καυσίμων, από τις οικοδομές κλπ. Άρα είναι πολύ ευεργετικό το αποτέλεσμα για τι ευρωπαϊκέ οικονομίε, Άλλωστε βοηθεί και στη δημιουργία εκατομμυρίων θέσεων απασχολήσεως στην Ευρώπη. Η ενεργειακή και κλιματική πολιτική της Ευρώπης, μέσα στο πλαίσιο αυτό δηλαδή, πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι ομοχλός για την ανάπτυξη. Και αυτά θα απορρεύσουν από τους στόχους. Όταν μιλούμε για στόχους της ενεργειακής αποδοτικότητας και όταν μιλούμε και για τη νέα οδηγία ενεργειακής απόδοσης που θα ε, υποβληθεί στο Κοινοβούλιο σύντομα, πιστεύω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να επιμείνουμε σε στόχους, σε θέσπιση στόχων. Χωρίς στόχους ενεργειακής απόδοσης δεν θα υπάρξει ανάπτυξη στην αποδοτικότητα της ενέργειας. Τέλος, χρηματοδότηση για τα μέτρα απόδοσης Ενεργειακή απόδοση για επενδύσει, δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι όμω μόνο το θέμα του ποσού των χρημάτων που θα δαπανίσουμε σε επενδύσεις αυτέ, Είναι κυρίως το πώς θα τα δαπανίσουμε, σε ποιο πλαίσιο θα δαπανίσουμε τα χρήματα, τα χρήματα αυτά. Πώς και ποιοι θα είναι αυτοί που θα υποφεληθούν από τις χρηματοδοτήσεις αυτέ. Μάλιστα, σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει και ο κύριος ε, Ζιλουάγκα. Ε, ε, Σας ευχαριστώ. Κατά την άποψή μας, ε, ο στόχος της ελληνικής αποδόσης είναι σημαντικός για δύο λόγους. Πρώτον, όπως ελέγχθη, σημαίνει ενεργειακή αποταμίευση περιβαλλοντική. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ σημαντική ποσόστοση μέσω των συστημάτων ε, θέρμανσης και ψήξης των κτηριακών. Άρα συνεισφέρουν αυτά στην κλιματική αλλαγή. Επίσης, η καλύτερη ενεργειακή απόδοση σημαίνει χαμηλότερη κατανάλωση από τα νοικοκυριά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας. Και μιλούμε για άνω του 10% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν μπορεί να διατηρήσει σε επαρκή θερμοκρασία το σπίτι του. Υπό την έννοια αυτή λυπούμεθα που τα κράτη-μέλη δεν έχουν τηρήσει τις ε, υποχρεώσεις ε, της οδηγίας, γιατί σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους, το 2020 θα είμαστε στην αποταμίευση του 18 με 19% ε, αντί για το 20%, αλλά σύμφωνα με μια μελέτη της Coalition for Energy Savings, κάποια κράτη-μέλη έχουν υπερβάλλει στην επίπτωση της νομοθεσίας τους για τα πρότυπα τακτηριακά. Εμείς θα θέλαμε να έχουμε δεσμευτικούς και συγκεκριμένους στόχους όπως ετήσια, ε, ετήσια ποσόστοση για την ε, ανακαίνιση των κτηρίων όπως λέγει το άρθρο 5. Επίσης θα πρέπει να υπογραμμίζουμε περισσότερο την, ε, το ρόλο της ενεργειακής απόδοσης ώστε να έχουμε ελάττωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Πρέπει να ελαττώσουμε την κατανάλωση ενέργειας στη συνολική μας, πέραν του να είμαστε πιο αποδοτικοί. Και για την απόδοση ως όφελος για τα νοικοκυριά, οι ανακαινήσει θα πρέπει να γίνουν με κοινωνικό χαρακτήρα, όπως λέγει το άρθρο 7, και ως καταπολέμηση ας πούμε, ε, ακριβώς της νεακής παινίας. Και δημοσιονομικώς μιλώντας, θεωρούμε ότι το επίπεδο των επενδύσεων δύσκολο θα μπορέσουν να καλύψουν την ταχύτατη μετάβαση προς ένα ε, ε, πιο βιώσιμο πρότυπο μοντέλο ενεργειακό. Και θα πρέπει να απευθυνόμαστε ε, στην, στους τελικούς πολίτες. Γιατί τελικώς εδώ μετατρέπουμε τους δημόσιους πόρους σε εγγυήσεις για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην πραγματικότητα. Και λέω, μια και έχουμε εκπρόσωπο της Κομισιόν, ότι βλέπουμε Διακόπτει ο Πρόεδρος. Κύριε Φιλουάγα, έχετε ολοκληρώσει το χρόνο σας. Ναι, ναι, τελειώνω. Δεν έχω τελειώσει ακόμα. Ε, για τις αναλύσεις κόστος ωφέλους δεν έχουμε καταλάβει το λόγο και ούτε η οδηγία το εξηγεί. Αν μπορούσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν να μας το εξηγήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σταμπουράνο. Συνάδελφοι, καλημέρα. Εμείς συμφωνούμε ότι πρέπει να απλουστεύσουμε και να επιταχύνουμε όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες οποιασδήποτε παρέμβασης και ιδιαίτερα μιλώντας για την ενιακή απόδοση. Εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι χρειαζόμαστε δεσμευτικούς στόχους η υποτένεια ότι θεωρούμε ότι δεν φτάνουν οι δηλώσεις και οι υποσχέσεις. Χρειάζονται στόχοι δεσμευτικοί στο 40%. Εάν κάποια κράτη-μέλη δυσκολεύονται να επιτύχουν τους στόχους αυτούς, αυτό δεν είναι αναγκαστικά συνέπεια του γεγονότος ότι έχουμε θέσει υπερβολικά υψηλούς στόχους. Θα έπρεπε να πάμε κράτος προς κράτος και να δούμε για ποιους λόγους ακριβώς κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτυχάνουν αποτελέσματα και άλλες όχι. Δεν θεωρούμε ότι είναι δυνατόν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουμε δύο, τρεις ή τέσσερις διαφορετικές ταχύτητες στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Και ούτε θεωρούμε πως μπορούμε να αφήνουμε πίσω κάποια κράτη-μέλη όπως να αφήσουμε πίσω κάποιον Ευρωπαίο πολίτη. Ε, Επανέχω λοιπόν ακριβώς στους πολίτες. Όλες οι παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, μικρής ή μεγάλης κλίμακος, είναι η καλύτερη επένδυση που ο μονομένος πολίτης και τα κράτη μπορούν να κάνουν για το μέλλον τους. Γιατί είναι επενδύσει που απέναντι στην διακύμανση των ενεργειακών αγορών είναι εγγυημένε επενδύσει, εγγυημένε από τους θεμελιώδεις νόμους θερμοδυναμικής, οι οποίοι υπερισχύουν των αγορών. Δεν υπάρχει καλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στις μελλοντικέ γενναίες από το να καταστήσουμε την Ευρώπη πραγματικά πιο δεκτική. Κάθε κιλοβατόρα που αγοράζουμε από το εξωτερικό, κάθε βαρέλι πετρέλαιο, κάθε κυβικό μέτρο φυσικού αερίου σημαίνει απορροή, έξοδο πλούτου προς τις χώρες από τις οποίες προέρχονται όλα αυτά και που πολύ συχνά αντιμάχονται των αρχών και των συμφερόντων μας. Επομένως η συζήτηση για την ενέργεια δεν είναι μόνο κλιματική και περιβαλλοντική. Δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά είναι και μια συζήτηση που έχει σχέση και με την ελευθερία και την δικαιοσύνη για τι μελλοντικέ γενναίε. Ευχαριστώ. Να σα υπενθυμίσω ότι θα έχουμε όλη την άνεση να συζητήσουμε αυτή την έκθεση και στη συνάντηση του Μαρτίου της Επιτροπής Ήτρε. Ας περάσουμε τώρα ε, στις ερωτήσεις των ομονωμένων ε, μελών. Να κλείσει τώρα ο κατάλογος μελετών. Και πλέον ε, όλοι οι θα έχουν ένα λεπτό στη διάθεσή τους και να σας ενημερώσω ότι θα είμαι και πιο αυστηρός από ότι προηγουμένως με τους κοιόδης. Παρακαλώ λοιπόν να τηρείτε το χρονικό όριο. Η κυρία Ροδρίγες. Gracias, presidente. Primero quiero señalar que Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλώ εκ μέρους της κυρίας Σολεδάθ Καβεθών, που είναι υπεύθυνη για το θέμα αυτό στην ΕΝΒΗ. Καταρχά να εκφράσω την δυσαρέσκειά μας που τα κράτη-μέλη δεν έχουν σταθεί στο ύψος των υποχρεώσεών του και δεν θα επιτύχουμε τελικά το 20%. Είναι αλήθεια βεβαίω ότι μαθαίνουμε από τα όσα συμβαίνουν και έχουμε σημειώσει τις δυσκολίες της αξιολόγησης και πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να μεταφράσουμε αυτή την εμπειρία, αυτή την εμπειρία σε πράξη. Για την επανεξέταση της οδηγίας ε, ενεργικής απόδοσης, εμείς θα προτείναμε να έχουμε μηχανισμός, μηχανισμούς που να βελτιώνουν τις, ε, τις συνθήκες ε, επενδύσεων στο πλαίσιο της ενεργικής απόδοσης. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τις στρατηγικές ανανέωσης, ανακαίνησης, με φύλλα πορεία εθνικά, οδικού χάρτες εθνικούς, με, όλους, ε, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Πρέπει να γνωρίζουμε ποια κτίρια πρέπει να υποστούν ανακαίνιση. Θα πρέπει όλες οι υποδομές του δημοσίου να προσυπογράφουν τι ε, υποχρεώσει αυτέ. Θα πρέπει τα αποτελέσματα της ε, παρακολούθησης και του ελέγχου που διεξάγονται υπό την οδηγία να σημειώνονται και να γίνονται δεσμευτικοί στόχοι. Σας ευχαριστούμε, διακόπτει ο Πρόεδρος. Και μία ερώτηση όμως, μία ερώτηση έχω για τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Έχετε αξιολογήσει την, τον αντίκτυπο των ε, μέτρων των κρατών μελών για την ε, αντιμετώπιση της νεακής παινίας ε, στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Μπένσον. Κύριος Μπένσον. Ευχαριστώ. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε μια κανονικά αποδοτική μετάβαση του ευρωπαϊκού συστήματο ενέργεια προ ένα μέλλον, ε, μια μελλοντική κοινωνία χαμηλή κατανάλωση άνθρακα. Είναι επίση να διασφαλίσουμε την εκπλήρωση των ενδεικτικών στόχων σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση με βελτίωση τουλάχιστον 27% βελτίωση τη ενεργειακή αποδοτικότητα μέχρι το 2030. Πρέπει να πετύχουμε του στόχου μα με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Ένα από τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα είναι το καθεστώ ε, υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά την αγική απόδοση, το άρθρο 7. Ανέφερε το 1% η Κομισιόν, αλλά ξέρουμε ότι παρέχονται 2 τρίτα των ε, γενικών εξοικονομήσεων ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να συμφωνεί και η Κομισιόν ότι αυτό το μέσο είναι απαραίτητο και αποτελεσματικό και για την επόμενη περίοδο. Και η χρηματοδότηση είναι σημαντική. Είναι δύσκολο αυτό το τομέα και από τη χώρα μου ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ε, με καρπούς που εύκολα θα μπορούσαμε να δρέψουμε, αλλά είναι χαμηλή η χρηματοδότηση. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει και αυτός, ε, αυτό το σκεπτικό, λαμβάνεται υπόψη. Ο κύριος Γκίρεκ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι κάναμε λάθος στην αρχή όταν υιοθετήσαμε αυτή την οδηγία. Γνωρίζαμε ευθύ εξ αρχής ότι η Ευρώπη ε, που δεν είναι ομοιόμορφη. Υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που είναι πιο εξελιγμένε και ανεπτυγμένε και κάποιες λιγότερο. Δεν μπορούμε λοιπόν με τον ίδιο τρόπο να αντιμετωπίσουμε τη μείωση κατά 20%. Ο δείκτης ήταν λανθασμένος ο δείκτης θα πρέπει να περιλαμβάνει και το κατακεφαλήν ΑΕΠ για κάθε κρατός μέλος. Μόνο τότε μπορούμε να εξετάσουμε την πραγματική αποδοτικότητα και όχι μόνο ε, την αριθμητική. Ε, γιατί για τις χώρες που θέλουν να αναπτυχθούν δεν μπορούν να ακολουθήσουν στους ίδιους ρυθμούς και να πετύχουν αυτό το 20% εξοικονόμηση. Και σας ρωτώ, ποιος θα είναι ο υπολογισμός για την Πολωνία πώς θα υπολογιστεί αυτός ο δείκτης ε, για την Πολωνία. Ο κύριος Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος. Όμως ε, το 2014 ήδη και στη δική μας Επιτροπή συζητήσαμε την κατάσταση σε έξι κρατημέλη και είδαμε ότι έχουν γίνει πολλές επενδύσεις σε αυτά τα κράτη-μέλη. Όμως ε, τα αποτελέσματα των επενδύσεων αναμένονται εντός των επόμενων 100 έως 300 ετών. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν όχι μόνο σε εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και μέτρα που θα συμβάλλουν στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Αλλιώς, απλώς θα πούμε ότι δεν έχει υπάρξει ε, σωστή χρησιμοποίηση και αξιοποίηση αυτών των κονδυλίων. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχα την τιμή να εκπροσωπήσω το Κοινοβούλιο στο Παρίσι και σε έτσι συμφωνώ με τις παρατηρήσεις πολλών μελών ότι πρέπει να ενισχύσουμε και όχι να περιορίσουμε ε, τις δεσμεύσεις μας, ιδίως σε ό,τι αφορά τα κτίρια. Είναι μία ε, άπαξ ε, δαπάνη και μετά όταν γίνει αυτή η επένδυση μετά περιορίζεται και περιορίζεται η επιπτώση του περιβάλλον και η ενεργική κατανάλωση. Πρέπει λοιπόν να το λαμβάνουμε αυτό υπόψη. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τα όσα είπε ο συνάδελφο ε, Μάρκο Πίπερο, συζητητή. Ανέφερε το ζήτημα των αλληλεπικαλύψεων. Θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει στα σχόλια του κύριου Πίπερ για τις αλληλεπικαλύψεις και ε, αυτό από μόνο του αυξάνει τη γραφειοκρατία και το κόστος. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω μια απάντηση προς αυτό. Ευχαριστώ τον κύριο Κέλλη. Ο κύριος Κάρινς. Ευχαριστώ πολύ. Έχω ορισμένε ερωτήσει προ την Επιτροπή. Δεν θέλω ε, να τοποθετηθώ. Ερωτήσει μόνο έχω. Περιορίζουμε λοιπόν τι εκπομπέ του του άνθρακα και καταλαβαίνω και αυτό που είπατε εσεί. Από ό,τι φαίνεται βρισκόμαστε εντό τροχιά για να πετύχουμε του στόχου μα. Το θέμα είναι τώρα η ενεργειακή αποδοτικότητα στην νομοθεσία σε ποιο βαθμό σχετίζεται με την μείωση των εκπομπών διοξιδίων του άνθρακα και σε ποιο βαθμό μα επηρεάζουν οι τεχνολογικέ εξελίξει ή η οικονομική επιβράδυνση. Η νομοθεσία είναι το πιο σημαντικό και σε ποιο βαθμό συμβάλλει στην γενικότερη κατάσταση. Σα ευχαριστώ που τηρήσατε και το χρονικό όριο. Ο κύριος Έριξον. Ευχαριστώ αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζει και η ε, κατάσταση στα ενεργειακά και στην ενεργειακή αγορά. Ξέρουμε ότι ε, υπάρχουν πολλές δυνατότητες από πλευράς ε, ενεργειακής απόδοσης και στα κτίρια. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι ενεργειακές τιμές πέφτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, κατά πιθανότητα προσωρινά βέβαια, πώς αυτό επηρεάζει και την οδηγία ενεργειακής απόδοσης. Είναι σημαντικό να το συζητήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλύσει πώς αυτό ε, θα αλλάξει και την, ε, τις επιπτώσεις και τον αντίκτυπο της οδηγίας. Και αυτό τι θα σημαίνει για μας. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την οδηγία ενεργειακής απόδοσης για να πετύχουμε τους ίδιους στόχους ε, βραχυπρόθεσμα. Ποιε θα είναι οι προεκτάσεις για μας. Ευχαριστώ. Τρομερή πειθαρχία επιδεικνύεται στο τέλος της συζήτηση. Και σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μάλλον βέβαια χρειάζομαι πριν ένα λεπτό, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Ο κύριος Πόλφερ και κύριε Καλνιέ και Πέτερσεν, αναφέρθηκαν ε, στο ζήτημα των κτηρίων. Να σας αναφέρω ότι θα έχουμε και μία αναθεώρηση της ε, οδηγίας ε, ακριβώς για αυτό το ζήτημα. Επομένω, ε, είναι σημαντικά τα κτίρια και για εμάς σε τη φορά την εξοικονόμηση ενέργειας. Ο κύριος Κάριντς ρώτησε τι βαθμό συνδέεται η ενεργειακή απόδοση με την μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Μέχρι τώρα δεν είναι ο βασικό παράγοντα βελτίωση. Προ το παρόν, η μετάβαση ε, στην, ε, σε μια κοινωνία χαμηλή ε, κατανάλωση άνθρακα έχει μεγαλύτερο αντίκτυο από ότι οι μετακινήσεις και οι αλλαγές σε τη φατινογική απόδοση. Στην επόμενη δεκαετία όμως θα δούμε ότι κάπως θα ισορροπήσουν τα πράγματα. Όμως αυτό συνδέεται και με τα μέτρα που θα λάβουν ε, τα κάτι μελη Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ωφέλη, και επανέρχομαι στα όσα είπε ο κ. Πέντερσεν, αν δεν μας ενδιέφερε το, το περιβάλλον και ότι το Παρίσι ήταν πολύ σημαντικό, το οποίο εμείς πιστεύουμε, και πάλι θεωρούμε ότι πρέπει να κινηθούμε προς την ενεργική απόδοση. Σίγουρα και στο ΑΕΠ είναι θετικός αντίκτυπος και στην απασχόληση. Ε, το φυσικό αέριο δεν ε, ε, δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας και μάλιστα δημιουργεί και εξάρτηση από τις χώρες εξαγωγούς. Υπάρχουν σαφή ωφέλη λοιπόν από πλευράς οικονομίας και σε ενεργειακού ανεφοδιασμού πέραν των υπολείπων. Είναι λοιπόν και οικονομική πολιτική, δεν είναι μόνο περιβαλλοντική. Μετά, τα όσα ανέφεραν ο κύριος Μπέντσεν και Γιάβορ, που είναι η χρηματοδότηση. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο κατά πόσο αυτέ οι επενδύσει έχουν νόημα, αλλά πώ θα λάβουμε αυτή την πρώτερη χρηματοδότηση για να γίνουν αυτέ οι επενδύσει Και έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να εξετάσουμε την καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων. Αναφέρθηκε λοιπόν ότι δεν πρέπει να γίνεται κατασπατάληση ή κακή χρήση αυτών των κονδυλίων και από την ε, πρωτοβουλία για τα FEE e κτίρια. Ε, ερχόμαστε σε επαφή ακόμα και με τις επενδύσει και με τις τράπεζε για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Αλλά πώς μπορούμε να βρούμε την πρώτη χρηματοδότηση στον κλάδο. Αυτό συνδέεται με την ε, συσσόρευση έργων αν θέλετε. Θέλουμε λοιπόν και τη γνώμη του Κοινοβουλίου για αυτά τα ζητήματα. Ο κύριος Φόχερ Ζιλβάγκερ και η κυρία Ροντρίγκες αναφέρθηκαν στο θέμα της ενεργειακής ένδυας. Η κυρία Ροντρίγκε μα ρώτησε ρητά αν έχουμε αξιολογήσει τον αντίκτυπο στην ενεργειακή ένδυα. Δεν έχουμε ακόμα αποτελέσματα, αλλά πρέπει να εξετάσουμε αυτό το τομέα. Δεν θα πω κάτι παραπάνω επ' αυτού. Και είναι ένα τομέα όπου ενδεχομένω η αναθεώρηση τη οδηγία να συμβάλλει περισσότερο. Είναι σύνθετο το ζήτημα, δεν είναι απλό. Όμω το εξετάζουμε στην αναθεώρησή μα και αν το Κοινοβούλιο και πάλι έχει σχόλια ή προτάσει, με τα χαρά να τα ακούσουμε. Ο κύριο Έριξον ζήτησε, με ρώτησε τι γίνεται με την τιμή του πετρελαίου. Δεν είναι η πρώτα απ' όλα ανταπόκριση στι αλλαγέ ζήτηση στην Ευρώπη. Όμω, πράγματι, αν συνεχίσουμε την πολιτική αυτή, θα μειωθεί και η ζήτηση ε, των καυσίμων. Δεν έχει νόημα λοιπόν να κάνουμε αυτή την πολιτική αν αυτό ε, απαιτεί ψηλέ τιμέ για να λειτουργήσει. Σίγουρα η τιμή είναι ο κύριο παράγοντα που οδηγεί τον κόσμο να λαμβάνει αποφάσει. Αλλά είναι ευρύτερο το ζήτημα. Ακόμα και στι ε, μεταφορέ, ε, στα κτίρια, στι επιχειρήσει δεν γίνονται πολλέ επενδύσει. Παρότι αυτέ οι επενδύσει θα είχαν. Ε, αποσβεστεί μέσα σε ένα χρόνο. Παρ' όλα αυτά δεν τις κάνουν. Η τιμή λοιπόν είναι πολύ σημαντικό παράγοντας, αλλά δεν είναι και τόσο καθοριστικό όσο σε άλλους τομείς. Ε, για τα πυρηνικά εργοστάσια δεν ε, έχω την απάντηση, θα έρθω σε επαφή με του συναδέλφου μου και θα του το μεταφέρω. Κύριο κύριος Κέλλη ανέφερε ότι δεν απάντησα ένα από τα σχόλια του κυρίου Πίπερ και ζητώ συγγνώμη γιατί ήθελα να επανέλθω σε αυτό για το ζήτημα των αλληλεπικαλύψεων. Δεν υπάρχει εκτίμηση ότι υπάρχει αλληλεπικάλυψη μεταξύ τη νομοθεσία και ενεργειακή απόδοση. Λοιπόν, για να το αναφέρω λοιπόν ρητό, έχουμε δύο ε, νομοθετικέ προτάσει για τα ελάχιστα πρότυπα ε, των πληροφοριών προ του καταναλωτέ. Έχουμε μία νομοθετική πρόταση για τα κτίρια που και πάλι θέτει ελάχιστα πρότυπα και δίνει στοιχεία και πληροφορίε στου καταναλωτέ. Έχουμε την οδηγία ενεργειακή απόδοση που αυξάνει τη ζήτηση για καλά προϊόντα και καλά κτίρια. Και έτσι συμπληρώνει τις πιο λεπτομερείς τεχνικές ε, νομοθετικές πράξεις που είναι πολύ σημαντικές με μια πιο οικονομική προσέγγιση και από πλευράς ζήτησης και από πλευράς ε, παροχής, προσφοράς ε, για να αντιμετωπίσουμε την αυξανόμενη ζήτηση αυτών των καλύτερων προϊόντων και κτηρίων δεν απάντησα σε ό,τι αφορά την διασύνδεση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και πάλι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε σωστά. Αν το κάνουμε σωστά, τότε το κίνητρο ε, θα υπάρξει κίνητρο και για τους ίδιους τους πολίτες ε, να βάλουν, ας πούμε, ε, ηλιακούς συσσωρευτές στην οροφή τους και ούτω καθεξής. Θα συνδεθεί δηλαδή και ως κίνητρο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κάτι τελευταίο. Ο κύριος Ταμεράνο είπε γιατί κάποιες χώρες μπορούν, ε, βλέπουν ότι πετυχαίνουν ε, τα αποτελέσματα που θέλουν και κάποιες όχι. Δεν το γνωρίζουμε, αλλά δεν, σίγουρα δεν είναι επειδή κάποιες είναι πλούσιες και κάποιες όχι. Κάποιες χώρες τα πηγαίνουν καλύτερα σε όλη την Ευρώπη και στο βορρά και στο νότο και παντού. Υπάρχουν δυνατότητες, αλλά αυτό είναι ζήτημα σωστής διακυβέρνησης, ε, διοίκησης ε, και όχι μόνο πόρων. Και αυτό με φαίνει και πάλι στο ζήτημα του κυρίου Γκιούρεκ. Παρότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο στόχος μας είναι ε, καθαρή ποσότητα ενεργειακής εξοικονόμησης, πράγματι δηλαδή έχουμε σε απόλυτους όρους αυτόν τον στόχο, σε εθνικό επίπεδο τα κράτη-μέλη μπορούν να, να, τα, να ορίσουν πώς θα πετύχουν αυτό το στόχο με τον τρόπο που επιθυμούν. Και βλέπουμε ότι και στην Πολωνία και αλλού υπάρχει πολύ καλή οικονομική απόδοση και έτσι περιμέναμε να υπάρχει και ανώτερος στόχος περιβαλλοντικά. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους γιατί ξεκινήσαμε καθυστερημένα και κάπως ε, έχουμε αντισταθμίσει αυτή την καθυστέρηση. Η έκθεση αυτή θα αποτελεί το κείμενο εξέταση ε, και το Μάρτιο. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της μέσας διάταξης. Το Δεκέμβριο του 2015 η Μπέρεκ... διακόπτει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Πίπερ, συγγνώμη. Δεν είμαι τόσο πεπειραμένος ως ε, Πρόεδρος. Μην ανησυχείτε Πρόεδρε. Μου φάνηκαν πολύ ενδιαφέρουσε ορισμένε παρατηρήσει που είχαν σχέση με την αποδόμηση τη γραφειοκρατία. Ο ίδιο ο κ. Χότσον δέχτηκε ότι στο άρθρο 7 υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει να απλοποιηθούν. Αυτό το άκουσα με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Ωστόσο, πάλι δεν απαντήθηκε μια κέρια ερώτηση. Μάλιστα Ορισμένοι εδώ είπαν εάν επιβάλλουμε την ε, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης είμαστε και πιο ανθεκτικοί απέναντι σε ενεργειακές κρίσεις. Σωστό. Όμως υπάρχουν και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε ορισμένες μάλιστα έχουν περάσει και το 50% της συνολικής ενέργειας. Υπάρχουν πάροχοι ενέργειας που έχουν εξειδικευτεί στην ανανεώσιμη πηγή ενέργεια. Τώρα, ντε και καλά θα επιβάλλουμε περιορισμού σε αυτού. Μπορούν να αποφασίσουν οι χώρε μέλη εάν θα επιλέξουν ίσω κάποια άλλα συστήματα. Για μένα αυτό το ερώτημα δεν απαντήθηκε. Εάν δηλαδή οι οριζόντιες αυτές, ε, οι οριζόντιες περιορισμοί θα επιβληθούν σε όλους. Ε, στο μεταξύ έχουμε για παράδειγμα στις σκανδιναβικές χώρες flat rate κατά αποκοπή για, τις ε, για την κατανάλωση της ενέργειας βασισμένες σε, ενεργειακή, ε, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κάπου νομίζω ότι έχουμε αυτοπαγιδευτεί μέσα σε όλες αυτές τις ε, ε, εκθέσεις και νομοθεσίες που έχουμε από τις αρχές του 2000, τις αρχές δεκαετίας του 2000. Όλα αυτά τα σημαντικά θέματα, περιλαμβάνει σημαντικά θέματα βεβαίως η οδηγία περί ενεργειακής απόδοσης και έχουν πολλή ουσία. Όμως πρέπει να τα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τη γραφειοκρατία. Εκεί θα ήθελα να ε, ακούσω προτάσεις, κάποιο input δηλαδή, και από άλλους συναδέλφους. Μάλιστα, σας ευχαριστώ κύριε Πίπερ. Το Δεκέμβρη 2015 η Μπέρεκ, η Μπέρετς, δημοσίευσε τις απόψεις της για την μεταρρύθμιση των κανόνων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η Κομισιόν αναμένεται να υποβάλει προτάσεις τον Ιούνιο φέτος η Μπέρετς έχει, επιβάλει, έχει υποβάλει μάλλον και προτάσεις για τις υπηρεσίες over the top, OTT, καθώς και για άλλα σχετικά θέματα. Α, έχουμε λοιπόν πολλά θέματα να συζητήσουμε. Έχουμε σχεδιάσει μια, έχουμε προβλέψει μάλλον μια ώρα και 15 λεπτά και με μεγάλη χαρά υποδέχομαι τον ε, κύριο Εσβάλλερ που είναι και πρόεδρος της Μπέρεκ. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι αντιμετωπίζουμε αυτό τον κόσμο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αλλάζει ταχύτατα. Αυτή η ψηφιακή μεταρρύθμιση ήταν και στο επίκεντρο του Νταβός την προηγούμενη εβδομάδα. Πρόκειται για μια επαναστατική ε, αλλαγή του ε, νομοθετικού πλαισίου και που αποτελεί και την καρδιά του μελλοντικού μας στόχου της ε, ψηφιακής αδενίας αγοράς. Και εκεί παίζουμε και ένα σημαντικό ρόλο για την ε, περαιτέρω αυτή νομοθεσία. Αυτό είναι το ιστορικό. Ε, σε ενώπιση του ιστορικού αυτού χαίρομαι για την ευκαιρία που μου δίνεται σήμερα μετά και από την μεταρρύθμιση του πλαισίου που ε, έχει υποβάλει η Μπέρεκ και της οποίες ηγούμε ε, ως πρόεδρος φέτος. Η επόμενη διαφάνεια σας παρακαλώ. Αρχίζουμε με το γεγονός ότι το πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες είναι ο βασικός πυλώνας της στρατηγικής για την κεντρική ε, ψηφιακή αγορά και μάλιστα ε, σχετικό ψήφισμα ανέκρινε και το Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει τρει βασικούς στόχους. Βελτίωση της πρόσβασης καταναλωτών και επιχειρήσεων. Δεύτερο, προωθημένα, προχωρημένα και καινοτόμα ε, δίκτυα και υπηρεσίες. Και τέλος, αύξηση της ψηφιακή οικονομίας. Αυτή η αναθεώρηση τη Telecom έχει ως στόχο να φτιάξει τις σωστές συνθήκες για ισότιμο ανταγωνισμό και τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν είναι η διασύνδεση, καθολικές υπηρεσίες, ισότιμος ανταγωνισμός και προστασία του φάσματος και τέλος ο θεσμικός σχεδιασμός. Η πρόκληση της ε, διασύνδεσης στην, ή της συνδεσιμότητας σε όλη την Ευρώπη. Πώς θα αναπτυχθεί η υποδομή ευρέως φάσματος και ταχαίως ευρέως φάσματος ώστε ξεπεραστεί η ψηφιακή, το ψηφιακό χάσμα και τέλος το ταχύ ευρύ φάσμα να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καταναλωτών με τις απαραίτητες επενδύσεις. Να τονίσω τώρα και να συμφωνήσω απόλυτα με τις απόψεις του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι οι επενδύσεις στις στα υπερταχαία δίκτυα θα πρέπει να βασιστεί σε ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού ο υψηλός ανταγωνισμός συνδέεται και με υψηλό επίπεδο επενδύσεων και επομένως χαμηλές τιμές για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Η Μπέρετς θεωρεί ότι εδώ τρία στοιχεία πρέπει να παίξουν ρόλο. Ε, ρύθμιση και όπου είναι απαραίτητο απορρίθμιση που πρέπει να συμπληρώνεται με, την, με τις θεσπίσεις για την καθολική υπηρεσία και κρατικές ενισχύσεις όπου αυτό είναι απαραίτητο. Σε ό,τι αφορά τις νομοθετικές ρυθμίσεις είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι ο ανταγωνισμός οδηγεί σε επενδύσεις. Επανέρχομαι στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που λέει και αυτό το ίδιο πράγμα. Ότι δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία που να λένε ότι η ενοποίηση των operator θα οδηγήσει σε αυξημένη επένδυση. Έχοντας πει αυτό, να μην λησμονείτε ότι για την επίτευξη των στόχων διασυνδεσιμότητας διαφορετικές προκλήσεις, διαφορετικές χώρες, πρέπει να επιλέγεται η βέλτιστη τεχνική λύση και το βέλτιστο μοντέλο που θα εξαρτηθεί από τα χαρακτηριστικά των διαφόρων αγορών. Επομένως δεν υπάρχει one size fits all λύση. Χρειάζεται ευκαμψία και χρειάζεται η ευκαμψία αυτή για να στηριχτεί ο ανταγωνισμός που θα αποδώσει τις μορφές εκείνες που είναι πιο ε, προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά της κάθε αγοράς. Θα υπάρξει δυνατότητα να ενισχυθεί και να ανανεωθεί το ρυθμιστικό, η ρυθμιστική εργαλειοθήκη για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις ε, διαφορετικές συνθήκες των αγορών στις χώρες μέλη. Αλλάξτε διαφάνεια. Σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη καθολική υπηρεσία. Εδώ μια γενική παρατήρηση. Η καθολική υπηρεσία εξακολουθεί να παραμένει σημαντικό μέρος του πλαισίου, του ρυθμιστικού πλαισίου και εξασφαλίζει την προσβασιμότητα στις βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε όλους για να ενισχυθεί η κοινωνική συμπερίληψη και να αποφευθεί το, ψηφιακό χάσμα στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τις ε, τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγέ στις αγορές πρώτα πρέπει να αναρωτηθούμε, είναι, υπάρχει ανάγκη να επανεξεταστεί το πεδίο εφαρμογής των ε, διατάξεων. Πρέπει οι χώρες μέλη να διατηρήσουν την ευχέρεια να καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής των καθολικών υπηρεσιών που μπορεί και να εξελιχθεί διαφορετικά ανάλογα με τις, ε, με τις εξελίξεις της αγορές των διαφόρων χώρων μελών. Επίσης να μην λησμονούμε ότι ο στόχος της καθολικής υπηρεσίας και των σχετικών παρεμβάσεων είναι η προσφορά βασικών ελάχιστων υπηρεσιών σε, μια, σε κάποιο ποιοτικό επίπεδο. Βέβαια, η καθολική υπηρεσία μπορεί να συμβάλλει και στον στόχο της διασυνδεσιμότητας. Χρειάζεται ανάληψη δράσης για να αποφευθεί το ψηφιακό χάσμα και να μην είναι οι χώρες μέλη εκείνες οι οποίες θα θεσπίσουν τεχνικά χαρακτηριστικά της πρόσβασης στο ευρύ φάσμα. Τώρα, ο ανταγωνισμό σε ισότιμου όρου. Βασικό στοιχείο τη συζητήσεω, διότι προκύπτουν νέε υπηρεσίε, ιδίω αυτέ που λέγονται over the top και που ανταγωνίζονται τι υπηρεσίε των παραδοσιακών παρόχων τηλεπικοινωνιών. Δύο θέματα εδώ. Υπάρχει στρέβλωση των ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων παικτών. ω γενική παρατήρηση θα τονίσω ότι συμφωνώ απόλυτα την άποψη της Ευρωβουλής που εκφράστηκε στο ψήφισμα και που λέει ότι αυξήθηκαν οι ψηφιακές υπηρεσίες και έχει αυτό ωφελήσει τους καταναλωτές και έχει οδηγήσει σε βελτίωση των επενδύσεων στις υποδομές. Γι' αυτό η Μπέρεκ προτείνει μια προσεκτική και διαφοροποιημένη προσέγγιση στο θέμα αυτό σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Μπέρεκ μιλεί για υπηρεσίες OTT1 που ε, θα, μπορέσουν να υποκαταστήσουν υπηρεσίες όπως WhatsApp και άλλες. Και στα τέλη του Φεβρουαρίου θα έχουμε έγγραφο το οποίο θα περιλαμβάνει τις θέσεις μας. Δεύτερη ερώτηση, ποιες είναι οι επιλογές και προοπτικές για το θέμα. Η Μπέρεκ προτείνει μια νομική βάση που θα επιτρέπει στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να παρακολουθούν τις εξελίξεις των αγορών ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών και πέραν από τις κλασικές ηλεκτρονικές τηλεπικοινωνίες και για να αντιμετωπιστεί κάποια έλλειψη συνοχής μέσα στις ισχύουσες διατάξεις. Ίσως χρειάζεται λοιπόν εκεί να γίνει κάποια διασάφηση. Τέλος, για να αποφευθούν ενδεχόμενες γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις πρέπει να γίνει ένας, μια αξιολόγηση ανακανόνα, rule by rule, για να εξεταστεί ποιες διατάξεις είναι, εξακολουθούν να είναι απολύτως αναγκαίες. Επόμενη διαφάνεια. Σε αυτό, στο πλαίσιο της προστασίας του τελικού καταναλωτού, η Μπέρεκ θεωρεί ότι δύο ερωτήματα πρέπει εδώ να απαντηθούν. Χρειαζόμαστε γενικές ή sector-specific νομοθεσίες. Η Μπέρεκ θεωρεί ότι χρειάζεται μια ισορροπία ανάμεσα σε γενικές διατάξεις και σε ειδικές ανατομία διατάξεις. σε χρόνους, σε, στις εποχές αυτές ταχύτατων αλλαγών για να αποφευθεί και η νομοθετική επικάλυψη αλλά και οποιοδήποτε νομοθετικό κενό. Δεύτερο, θεωρούμε, έχουμε δηλαδή εδώ στη δεύτερη ερώτηση σχετικά με το επίπεδο εναρμόνισης του καταναλωτικού δικαίου. Η Μπέρεκ θεωρεί ότι οι χώρες μέλη και οι ρυθμιστές πρέπει να μπορούν να ανταπογκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών και να επιτρέπουν χώρο για ε, πειράματα με νέες τεχνολογικές λύσεις. Χρειάζεται λοιπόν καλύτερα αυτό παρά να είναι πλήρως εναρμονισμένες προσεγγίσεις. Εξάλλου, πλήρης εναρμόνιση εμπεριέχει κινδύνους και μπορεί να καταλήξουμε έτσι σε ελάχιστου κοινού παρονομαστές, το οποίο δεν επιθυμούμε. Επίσης, η Μπέρεκ γνωρίζει ότι το φάσμα είναι ένα από τα κέρια θέματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιτρέψτε μου λίγα λόγια σχετικά με το status quo. Σύμφωνα με την άποψη της Μπέρεκ, το υφιστάμενο πλαίσιο αποδίδει, λειτουργεί καλά και προσφέρει αξία στον καταναλωτή και προσφέρει τη δυνατότητα επενδύσεων και στα πλαίσια των νέων δικτύων τέταρτης γενναίας. Υπάρχει περισσότερος χώρος για τις νέες αυτές γενναίες στην Ευρώπη, όπως και αλλού, Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία, περισσότερο εδώ. Επίσης η εναρμόνιση που γίνεται στην Ευρώπη είναι πραγματικότητα. Οποιαδήποτε λοιπόν παρέμβαση, περαιτέρω εναρμόνιση θα πρέπει να εξεταστεί πρώτα πολύ προσεκτικά και να γίνει εξισορρόπηση, να γίνει στάθμιση ωφελών και επιβαρύνσεων. Οι στόχοι της διασυνδεσιμότητας και της ικανότητας φάσματος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τις υπηρεσίες και για την κατανομή φάσματος στις διάφορες χώρες μέλη. Στα πλαίσια αυτά, οποιαδήποτε άλλη εναρμόνιση εκ των άνω διατρέχει τον κίνδυνο να καταλήξει σε μία αποτελεσματική χρήση αυτής, αυτού του πόρου, του σπάνιου πόρου που είναι το φάσμα. Το εφιστάμενο πλαίσιο αναγνωρίζει ήδη και προσφέρει εργαλεία για εναρμόνιση του φάσματος των ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών και θέτει και χρονοδιαγράμματα για την επιβολή των ρυθμίσεων αυτών. Χρειαζόμαστε και ε, πιο στενή συνεργασία ανάμεσα στην ε, Radio Spectrum Policy Group και την BEREC. Μου αφήνετε να κάνω ακόμα μερικά σχόλια για τα σχέδιά μας, λέει ο πρόεδρο της BEREC στον πρόεδρο της Επιτροπής. Τελευταίο κρίσιμο θέμα είναι ε, ο θεσμικός σχεδιασμός. Γνωρίζετε ότι πάντοτε έχουμε επικριθεί σε ό,τι αφορά το θεσμικό σχεδιασμό. Εμείς θεωρούμε ωστόσο ότι η Μπέρεκ πρέπει να παραμείνει στον θεσμικό σχεδιασμό και θα πρέπει να επιμείνει σε αυτή την ε, θέσπιση στόχων για, σε συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές για την αποτελεσματικότητα του έργου της Μπέρεκ. Ωστόσο, ο θεσμικός σχεδιασμός θα πρέπει να παραμείνει ως έχει. Αυτό πιστεύουμε εμείς. Ε, η τελευταία μου διαφάνεια δείχνει για την συνέχεια που δίνεται στο TSM. Βλέπετε στην διαφάνεια αυτή ότι μας μένει πολύ δουλειά να κάνουμε ακόμη αφενός για την ουδετερότητα του δικτύου. Εκεί επεξεργαζόμαστε κατευθυντήρες γραμμές και στα τέλη του Αυγούστου θα έχουμε κάποια, ε, κάποιες προτάσεις. Συζητούμε επίσης για την περιαγωγή, το roaming. Αυτή είναι η στόχη της Μπέρε και σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ε, Σα ευχαριστώ. Οι σκιώδει εισηγητέ ε, τώρα παρακαλώ. Δύο λεπτά έκαστο. Ευχαριστώ κυρία Νίμπλερ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Εσφάιλερ για τα όσα εξηγήσατε. Πρώτο ένα σχόλιο. Σα υποστηρίζω απόλυτα ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι επενδύσει, ιδίω για το ε, υπερταχή φάσμα χρειάζεται να δώσουμε κίνητρα όπου αυτό είναι δυνατό. Σα υποστηρίζω απολύτω. Αν θέλουμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη, το α και το ω είναι να ενισχύσουμε την ε, ρακοκαλιά του δικτύου μας προσφέροντας το ταχύ φάσμα όσο, όπου αυτό είναι δυνατό. Ερώτηση πρώτη. Πολιτική συχνοτήτων. Είπατε, εγώ μάλλον θα ήθελα να είμαι λίγο πιο προοδευτική και να ρίξω μια ματιά στις εφαρμογές από, την αυτο, από τα αυτόματα αυτοκίνητα που δημιουργούνται αυτόματα δηλαδή μέχρι την προσφορά υπηρεσιών υγείας από το διαδίκτυο μέχρι το διαδίκτυο 4.0 χρειαζόμαστε εκεί σημαντικά βήματα εναρμόνισης μέχρι που θα θέλατε να φτάσετε εκεί θα ήθελα επίσης να δω και αν γίνεται κατανοητή ανάγκη μια συνολικής ευρωπαϊκής προσέγγισης τώρα δεύτερο ουδετερότητα διαδικτύου και είναι οι δικέ από την πράξη. Υπάρχουν παράπονα καταγγελίες. Τελευταίο, ίση όρια ανταγωνισμού. Μπορείτε να εξηγήσετε κάπως περισσότερο. Πού διαπιστώνετε ότι λόγω των διαφορετικών κανόνων παιχνιδιού οδηγούμαστε σε κάποιες τρευλώσεις του ανταγωνισμού και τι μπορούμε να κάνουμε με την εργαλειοθήκη που διαθέτουμε. Θα αρκεστώ σε αυτά και κύριε Πρόεδρε τήρησα το χρόνο αγόρευσης. Πολύ καλά. Μπράβο σας κύριε Νίμπλερ. Η ε, κυρία Κρέλ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομη παρατήρηση, δύο ερωτήσεις. Βεβαίως η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η υποδομή. Είμαι βεβαία ότι εκεί μένουν πολλά να γίνουν ακόμη. Όχι μόνο αν θα χρησιμοποιήσουμε κρατικές ενισχύσεις εκεί ε, ή αν θα οργανώσουμε τον ανταγωνισμό με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστεί δυνατόν να υπάρξουν διαφορετικά μοντέλα ε, αγορών τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Δεύτερο, η οργάνωση της ψηφιακή ενίας αγοράς που είναι και το μεγαλύτερο εργοτάξιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φέτος. Επ' αυτού το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο στην έκθεσή του για την ψηφιακή ενία αγορά είπε ότι θα πρέπει να αποδοθεί ενισχυμένο ρόλο στην ΠΕΡΕΚ στην εργασία αυτή. Θέλουμε να δώσουμε ισχυρότερες αρμοδιότητες στην ΠΕΡΕΚ. Κυρία Σβάιλερ, τι θα θέλατε να δείτε εσείς. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή ώστε να βελτιωθεί η εργασία και η συνεργασία. Εγώ με την ΠΕΡΕΚ έχω ως τώρα συνεργαστεί θαυμάσια και νομίζω ότι πραγματικά ως οργάνωση κάνετε καλή δουλειά. Το ερώτημα είναι επίσης πώς μπορεί να ενισχυθεί το γραφείο που διατηρεί η ΠΕΡΕΚ στην Ρήγα. Θα συμφωνήσω και με την κυρία Νίμπλερ για το θέμα της ουδετερότητας του δικτύου. Έχω την εντύπωση ότι διάφοροι ε, φορείς εξακολουθούν να έχουν διαφορετικές απόψεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε καθαρά τι πιστεύουμε εμείς για την ουδετερότητα του δικτύου. Συμφωνείτε εσείς με τα όσα είπαμε και με την έκδοση των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών για να μην μείνουμε και τελευταίοι σε όλη αυτή την προσπάθεια. Βλέπετε ότι τήρησα το χρόνο μου. Ευχαριστώ κυρία Κρέλ. Θαυμάσια λέει ο πρόεδρος. Ομάδα ECR, Κύριο Χένκελ. Κοιτάξτε, εγώ πέρασα όλη μου τη ζωή σε αυτή την ε, βιομηχανία και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους καθυστερούμε, είμαστε καθυστερημένοι εναντί των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν ότι προχωρήσαμε πολύ αργά στην ε, προσαρμογή της ε, νομοθεσίας σχετικά με τις κρατικές ε, επιχειρήσεις κυρίως. Η κυρία Κάλλας και με το ρυθμό των ιδιωτικοποίησεων. Έχω ε, κάποιες ερωτήσεις. Καταρχάς για το ισότιμο παιχνίδι στην OTT. Είπατε ότι αντίστοιχοι κανόνες πρέπει να ισχύουν για αντίστοιχες Συγκρίσιμε εν πάση περιπτώσει υπηρεσίες, αλλά πρέπει να καταλάβει κανείς ποιε είναι αυτές οι υπηρεσίες. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να διαφοροποιούμε μεταξύ της πρόσβασης στα δίκτυα και της πρόσβασης στις υπηρεσίες. Γιατί η πρόσβαση στα δίκτυα προφανώς χρειάζεται ρύθμιση για να έχουμε ανταγωνισμό στην αγορά. Αλλά οι υπηρεσίε και αυτέ μπορούν να τύχουν ρύθμισης. Επίσης μιλήσατε για εναρμόνιση. Και εκπλήσωμαι, διότι λέτε ότι πρέπει να προχωρήσουμε με προσοχή. Όταν μιλούμε για το διαδίκτυο των πραγμάτων και μιλούμε για ομοιογενή προσέγγιση για το φάσμα και, και αυτό εναρμόνιση δεν σημαίνει. Επίσης, για τον θεσμικό σας ε, σχεδιασμό. Μας λέτε ότι έχει λειτουργήσει πολύ καλά, αλλά η Μπέρεκ είναι ακόμα ένα σώμα 28 διαφορετικών ρυθμιστικών αρχών. Ε, τι θα γίνει λοιπόν με την ουδετερότητα του δικτύου, τι θα γίνει με την TSM που πρέπει να ισχύσει αντίστοιχα. Η Μπέρεκ θα προχωρήσει στη δουλειά αυτή και πώς θα χειρίζεστε την επίλυση διαφορών εφόσον υπάρχει δηλαδή η απόκληση μεταξύ των ρυθμιστών. Ευχαριστούμε κάλλας. Ε, εξαιρετικά τα πάμε με το χρόνο. Ο κύριος Ράιμοντ. Ευχαριστώ κύριε έσφαλε Μία ερώτηση. Σχετικά θεμελιώδης ερώτηση. Σεις, Μπέρεκ δηλαδή, αλλά και εσείς, πώς αντιδράτε από άποψη δημοκρατίας στις ε, εξελίξεις. Μιλάμε πολύ εδώ για προστασία καταναλωτών, αλλά ε, το διαδίκτυο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και δημοκρατικά. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να οριστεί η καθολική υπηρεσία. Δεν είναι μονάχα ζήτημα αγοράς. Το βάθρο πάνω στο οποίο στέκεται είναι η δημοκρατική πολιτική. Κατά πόσο παίζει αυτό ένα ρόλο στους μελλοντικού σχεδιασμούς σας. και πέραν από την ενατένιση των αγορών και των καταναλωτών. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ. Ας πάμε τώρα στις ε, ερωτήσεις. Ο κ. Ευχαριστώ. Πρώτα, η εισαγωγή του 5G, της πέμπτης γενεάς. 2020 δεν είναι κάπως αργά. 2018 είναι καλύτερα γιατί υπάρχει η Κορέα και η Ιαπωνία που είναι σχεδόν έτοιμες. Δεύτερο, εναρμόνιση για ολόκληρη την Ευρώπη. Χρειάζεται και εκεί θα εφόσον χρησιμοποιηθούν οι αποδόσεις των πληστηριασμών για επενδύσεις δεν θα είναι σημαντικό αυτό για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη ε, μιλείτε και συνεχίζετε και με την ίσο ISO δηλαδή για ε, την πρόθεση των θεμάτων αυτών και μία ερώτηση ακόμα η μέγιστη MTR. Ποια θα είναι η μέγιστη απόδοση της MTR. Κύριε Μπόνι, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την πλήρη παρουσίασή σας και την παρουσίαση του πλαισίου τηλεπικοινωνιών. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις επενδύσεις Και τι λέτε για αυτή, για αυτή την κοινή προσπάθεια με την Europe Facility, τα διαρθρωτικά ταμεία, τα περιφερειακά ταμεία και τα ε, ταμεία ευρωπαϊκής στρατηγικής. Επίσης, λέτε ότι είμαστε εν μέσω της διαδικασίας εναρμόνισης, αλλά σκεπτόμενοι την πέμπτη γενεά, το 5G, πρέπει να προετοιμάσουμε και το δικό μας ε, φύλλο πορείας προς το 5G σε συνεργασία με κάποιους διεθνείς φορείς και οργανισμούς αλλά τι λέτε για την εναρμόνιση στα πλαίσια του φύλου αυτού πορείας επίσης για τις ε, συνολικές υπηρεσίες είπατε ότι η επικαιροποίηση των κανόνων θα πρέπει να γίνει τις εθνικές κυβερνήσεις αλλά αν θέλουμε να αποφύγουμε κάποιες λύσεις που θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνες για την ευρωπαϊκή εναρμόνιση πώς θα δώσουμε και την αρμοδιότητα στις, κυβερν... στις εθνικές κυβερνήσεις διατηρώντας την αρμόνιση. Ευχαριστώ η κυρία Βαλέα. Σας ευχαριστώ. Μιλούμε για την ολοκλήρωση και τον ανταγωνισμό σαν να είναι εχθροί. Αλλά εάν η πρόσβαση δεν ενταχθεί πλήρως στο πλαίσιο, πώς αυτά τα δύο είναι στοιχεία που συγκρούονται. Λέτε ότι στο παρόν μοντέλο ακόμα εργαζόμεθα, αλλά χρειαζόμαστε επενδύσεις στις, στις υποδομές. Αλλά τι σημαίνει αυτό, έχουμε φτάσει σε ένα όριο κερδοφορίας που θα απέτρεπε περαιτέρω επενδύσεις αυτή τη στιγμή. Και αν είναι έτσι, τι χρειαζόμαστε ως παροχή κινήτρων για να πάμε στην επόμενη φάση της αγοράς. Ευχαριστούμε. Τελευταία ερώτηση, η κυρία Κούμπουλα Νάτρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η υψηλή ταχύτητα και η κάλυψή της θα πρέπει να είναι πρώτης προτεραιότητας για να μείνουμε σε επαφή με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ε, για μια νέα ηγετική θέση της Ευρώπης. Αλλά σχετικά με την ε, οδηγία για τις υπηρεσίες, τι θεωρεί η Μπέρεκ ότι είναι ακόμα επικαιροποιημένη, τα phone boxes τα χρειαζόμαστε ακόμα, χρειαζόμαστε τους τηλεφωνικούς καταλόγους, ε, τους τυπωμένους, τουλάχιστον εμείς στη Βιλανδία δεν τους πλέον. ή, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, αποστοχούν στην ε, συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας το οποίο προέκυψε και από το σεμινάριο που ε, διοργανώσαμε στο S&D σχετικά και με αυτούς που ψάχνουν να βρουν δουλειά και τις εμπορικές υπηρεσίες και τις δημόσιες υπηρεσίες υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις και πρέπει να ηγηθούμε ελπίζω ότι η Μπέρεκ κινείται ηγείται της προστασίας μαζί μας. Ε, και την ίδια ερώτηση για το 5G. Γιατί αυτή η επιφυλακτικότητα, αυτή η προσοχή με την οποία πρέπει να προχωρήσουμε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να τρέξουμε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βίλιαν. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Κοιτάξτε, εμείς ε, στην Κομισιόν έχουμε συνεργαστεί πολύ στενά με την Μπέρεκ. Η προηγούμενη γνωμοδότηση ήταν το αποτέλεσμα μιας μακράς ε, επίσημης και ανεπίσημης συνεργασίας και θα συνεχίσει μέχρι τη στιγμή που θα υποβάλουμε πρόταση στους συνομοθέτες και νομίζω ότι είχαμε πάρα πολλά σημεία συμφωνίας και σύγκλησης κατά τη διαδικασίας αυτής. Για να θίξω κάποια μόνο από τα θέματα που έθιξε και ο πρόεδρος και τα μέλη. Στη δημόσια διαβούλευση εντυπώσαμε ευρύτατη στήριξη για υψηλής ταχύτητας ε, συνδέσεις και καλή προσβασιμότητα στο σύνολο του ευρωαϊκού εδάφους. Αυτό εντοπίστηκε ως βασικός στόχος της αναθεώρησης του πλαισίου. Το πώς αυτό από εκεί πέρα ε, περνάει μέσα από τα διάφορα νομικά στοιχεία του πλαισίου ως προς την πρόσβαση στα δίκτυα και την ε, προώθηση του ανταγωνισμού ο Επίτροπος μόλις εκθέσει. Επιβεβαίωσε ότι ο ανταγωνισμός είναι βασικός μοχλός κίνησης των επενδύσεων αλλά βεβαίως σε ένα πνεύμα εργαλειοθήκης όπως είπε και ο κύριος Εσβάιλα πρέπει να δούμε κατά πόσον μπορούμε να εξοπλίσουμε το πλαίσιο με καλύτερα εργαλεία που θα μπορούσαν να υποστηρίζουν ακόμα καλύτερα τις επενδύσεις μέσω εναλλακτικών παρόχων αλλά και των κλασικών παρόχων. Δηλαδή όλοι να έχουν τις, ε, την ευκαιρία να αντλήσουν ωφέλειες από τις ε, πρόσθετες επενδύσεις που επιθυμούν όλοι να συμβούν. Καλύτερη πρόσβαση και στην ε, νομοθεσία επομένως μέσω της βελτίωσης των υποδομών και των δικτύων. Για το θέμα του φάσματος Εμείς το υπογραμμίζουμε πάντοτε αυτό το ζήτημα με ισχυρότατες πλειοψηφίες ψηφίσατε εδώ για τον συντονισμό της χρήσης του βάσματος στους τελευταίους μήνες της προηγούμενης εντολής του Ευρωκοινοβουλίου και το οποίο ήταν σημαντικότατο πολιτικό θέμα της ταυτοποίησης δηλαδή των πιο σημαντικών περιοχών της αναθεώρησης του πλαισίου για το φάσμα. Και εμείς θεωρούμε ότι, όπως είπε και ο κύριος Σέσβάιλα, ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα η εναρμόνιση του φάσματος να προχωρήσει για τις υψηλής ταχύτητας τηλεπικοινωνίες, όπως το 5G, και την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο για, το, για τη δέσμη των 500, αλλά έχουμε ομόφωνες τοποθετήσεις από τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το πώς διατίθεται το φάσμα στους παρόχους, το χρονοδιάγραμμα, τις, τις Συνολικά λοιπόν θα έλεγα ότι η κάλυψη των δικτύων που χρησιμοποιούν το φάσμα είναι πολύ σημαντική ε, ως συνολικός στόχος και, και στην ανάθεση συγκεκριμένων τμήματων του φάσματος και εθνικά. Ευχαριστούμε τον κύριο Βίλιαμ. Ο κύριος Έσουαϊλα τώρα έχετε λάβει μια σειρά από εξαιρετικές νομίζω ερωτήσεις και όλοι ελπίζουμε ότι θα λάβουμε και εξαιρετικές απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσουμε την κυρία Νίπλα και το ζήτημα της μεγαλύτερη εναρμόνιση της συχνότητας. Η Βέρα Γέννη συμφωνεί ότι το χρονοδιάγραμμα για την απολευθέρωση του φάσματος ε, από τις Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Επικοινωνιών είναι σημαντικό ζήτημα για την Ευρώπη, ιδίω ό,τι αφορά την ανάπτυξη του 5G. Είναι απολύτω σωστό αυτό που είπατε. Όμω, κατά τη γνώμη μα, η, κοινή, η μάλλον σημερινή διαδικασία εναρμόνιση του χρονοδιογράμματο ήταν πολύτιμη για την αγορά και για του τελικού χρήστε. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει τη δυνατότητα και την εξουσιοδότηση να, αποδεσ... να την αποδέσμευση του φάσματος εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Η εναρμόνιση του φάσματος ε, γενικώ πώς είναι σημαντική και σχετίζεται και βλέπουμε ότι γίνεται από την ITU γενικότερα, διεθνή οργανισμό με τον οποίο απονέμεται το φάσμα σε διαφόρου χρήστε, αλλά και από το CPT. Από αυτή την πλευρά λοιπόν χρειαζόμαστε μια πιο στενή συνεργασία από ευρωπαϊκή πλευρά εντό τη ε, ITU, CPT, BEREC και SPG. Όμως ε, πρέπει να δούμε πώ μετρούμε ακριβώ αυτό το καλύτερο συντονισμό. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει το πλεονέκτημα του ε, πρώτου. Το μάθαμε και στο ε, φάσμα των 700 MHz. Χώρες όπως η Γαλλία που ε, δίσταζαν να κάνουν αυτό το βήμα έμαθαν από όλη αυτή τη διαδικασία μέσω του συντονισμού ότι είναι καλή ιδέα να γίνονται αυτές τις θερμοπρασίες των 700 MHz. Γι' αυτό και η γαλλική διοίκηση αποφάσισε να μας ακολουθήσει. Βρισκόμαστε στην αρχή των διαπραγματεύσεων, όμω θεωρούμε ότι η Μπέρεκ έχει δίκιο ως προς αυτό. Τώρα, στην ουδετερότητα του δικτύου. Ξέρετε ότι θα υπάρξει και ένα εσωτερικό εργαστήριο κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας μας ε, στο Ρότερνταμ. Θα προσκαλέσουμε εκπροσώπους του ακαδημαϊκού χώρου για να δούμε ποιες προτάσεις έχουμε στη διάθεσή μας, θα αναλύσουμε την ε, εντολή FCC για την ουδετερότητα του δικτύου και υπάρχει εδώ όντως ένα ζήτημα. Πρέπει να καταλήξουμε σε κρατητήρες γραμμές του πλευράς Μπέρεκ για να καταδείξουμε ότι υπάρχει βούληση να προχωρήσουμε αυτή τη διαδικασία με συγκεκριμένες προτάσεις. Και για το θέμα του OTT το εξετάζουμε κατά κανόνα. Εξετάζουμε το ζήτημα ε, του ίσου πεδίου ανταγωνισμού, αν είναι ζήτημα ρυθμιστικού πλαισίου ή αν είναι θέμα προστασία δεδομένων, θέματα ασφαλείας. Εντός της Ομοσπονδιακής αυτής αρχής πήραμε μια απόφαση για το Gmail της Google, ότι πρέπει δηλαδή να πληρεί τις ίδιε υποχρεώσεις, όπως ε, οποιοδήποτε άλλη υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Διεξάγεται λοιπόν μια νομική συζήτηση για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Γιατί στη Γερμανία αυτό έχει φτάσει μέχρι επίπεδο διοικητικού δικαστηρίου. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποια θα υπάρξει μια διαδικασία εξέταση και διαπραγμάτευση στα νομικά ζητήματα. Τώρα την κυρία Κρέλ. Ποιο είναι ο θεσμικό σχεδιασμό, ποιε είναι οι επιθυμίε του Μπέρεκ. Θεωρούμε ότι υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο περιθώριο βελτίωσης, όμως εν γέννη αυτό το μοντέλο των δύο πυλώνων, ότι αφενός έχουμε την υπηρεσία της Μπέρεκ με τα κεντρικά της στη Ρήγα και εν γέννη ε, Μπέρεκ ω θεσμικό όργανο σου είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί και θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω εσύ μαζί με την ΒΕΡΕΚ αλλά και εσείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορείτε να δείτε και να αξιολογήσετε τη δουλειά που κάνει η ΒΕΡΕΚ. Ότι αναγνωρίζεται και από αλλού και από την FCC και από, άλλους, ε, από άλλες ρυθμιστικές αρχές. Έχει λοιπόν αποδείξει την αξία του αυτό το μοντέλο. Για το OTT. Έκανα κάποια σχόλια. Μετά. MTR. Κύριε Ρούβικ. Η πολιτική της ε, ορθής χρήσης και περιαγωγή. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς. Ξέρετε ότι το Ρευτήρι Βέρεκ ακόμα εξετάζει αυτό το θέμα. Είναι πολύ νωρίς όμως ε, να σας δώσω συγκεκριμένα στοιχεία. Και το θέμα του MTR ήταν κρίσιμη σημασία, όμως νομίζω θα βρούμε λύσεις από αυτού. Ε, το κύριο Μπόνι, το θέμα των ε, ταμείων. Είμαστε υπέρ της προσέγγισης ε, με γνώμονα την αγορά και τα ταμεία μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά. Όμως μας ενδιαφέρουν οι ιδιωτικές επενδύσεις στον κλάδο γιατί ο ανταγωνισμός και οι ιδιωτικές επενδύσεις κατά τη γνώμη μας είναι ο καλύτερος δρόμος. Νομίζω αυτά ήταν τα κύρια θέματα που θίξατε. Κύριε Χένκελ, Ναι, δεν απάντησα στο δικό σου ερώτημα. Ναι, είναι για μένα σημαντικό, λέει ο Πρόεδρο. Πολιτικό ζήτημα, αλλά έχει επιληθεί όχι από τι εθνικέ αρχέ. Αυτό θα πρέπει να το απευθύνεται στο Συμβούλιο των Υπουργών. Κάτι πολύ συγκεκριμένο ε, για την οδηγία περί δημοσίων υπηρεσιών, καθολικών υπηρεσιών. Μάλλον θα συμπεριληφθεί και στην πρόταση της Κομισιόν το καλοκαίρι. Είναι πολύ λοιπόν συγκεκριμένο το ερώτημά μου. Εκτός μικροφώνου. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Θα υπάρξει μια αναθεώρηση της οδηγίας αυτής. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Βρισκόμαστε στο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Ναι, νομίζω ότι έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματα. Ευχαριστούμε τον κύριο Έσβάιλα για την παρουσία του εδώ σήμερα, για την παρουσία που μας έκανε και για το ότι απάντησε σε όλες τις ε, ερωτήσεις. Και προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τα χαιρετίσματά μας στον κύριο Έτιγκερ. Κυρίε και κύριοι, επειδή ακριβώς ήμασταν τόσο πειθαρχημένοι στη συζήτηση, μπορούμε με άνεση χρόνου να περάσουμε στο επόμενο σημείο της μέσης διάταξης. Ε, ενημέρωση για τους ε, τριμερείς ε, διαλόγους. Η κυρία Δερκαστήγιο Βέρα δεν είναι εδώ σήμερα και πρέπει να επενθυμίσω ότι είναι η συγγήτρια της ιτρέ για την ε, οδηγία δικτύων και ασφάλεια πληροφοριών η ΙΤΡΕ είναι συνδεδεμένη επιτροπή υπό τον κανόνα 54 και η γνωμοδότηση υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο του 2013 στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Δεν είναι εδώ η κυρία Πιλάρ Δεκαστήγιο. Επομένως, μου ζήτησαν να συνοψίσω εξ ονόματός της τα κύρια απορίσματα. Είναι η πρώτη νομοθετική πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και είναι το πρώτο σημαντικό βήμα ε, προς, το, προς ψηλά επίπεδα ασφάλειας στο διαδίκτυο στην Ευρώπη. Η οδηγία θα κάνει τα εξής τρία πράγματα. Πρώτον, οι εμπορευόμενοι βασικών υποδομών, οι βασικοί πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να εφαρμόζουν ε, τεχνολογίες εχμής σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και να κοινοποιούν τυχόν ε, παραβάσεις και προβλήματα που συνδέονται στην ασφάλεια στις αρχές. Πρέπει να προσδιορίζουν αντίστοιχες στρατηγικές και να έχουν και αντίστοιχες ομάδες ανταπόκρισης για να αναλύουν και να παρακολουθούν απειλές και να ανταποκρίνονται σε επιθέσεις στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών από εδώ και πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή θα είναι σε καλύτερη θέση να ανταποκριθεί στις ε, συνεχείς απειλές στον κυβερνοχώρο και έτσι θα διαμορφώσουμε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας. Επί τη ευκαιρία ήθελα να συγχαρώ την κυρία Δελκαστήγιο για τα πολύ ε, σημαντικά επιτεύγματά της ε, και μας λέει ότι αν υπάρχουν ερωτήσεις βεβαίως μπορείτε να τις θέσετε, είναι ευπρόσδεκτε. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Κέλλη από πλευράς Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι τιμή μου για τον κανονισμό προστασίας δεδομένων να είμαι η συγκητής του ΕΛΚ είχε προταθεί από την Επιτροπή Reading το 12 επανήλθαμε το Φεβρουάριο του 2013 και το Μάρτιο του 2014 στην Ήτρε και τέλος υπό την Λετωνική Προεδρία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2015 το οποίο άνοιξε το δρόμο για τους ε, τριμερείς διαλόγους που ξεκίνησαν αμέσως υπό την ε, Προεδρία Λουξεμβούργου και μετά από εννέα τριλόγους συμφωνήσαμε το Δεκέμβριο του 2015. Και βεβαίως πρέπει να αναγνωρίσουμε εδώ τις προσπάθειες της ε, Λουξεμβουργιανής Προεδρίας για τον τρόπο με τον οποίο ηγήθηκαν, οδήγησαν αυτές τις συζητήσεις τους τριλόγους. Τώρα, Ελπίζω ότι η διάταξη αυτή θα παραμείνει για πολλά χρόνια. Αφενός είναι κανονισμός που σημαίνει ότι είναι πανευρωπαϊκός νόμος για την προστασία δεδομένων που αντικαθιστά τους 28 ή περισσότερους μέχρι στιγμής. Επίσης είναι ενιαία θηρίδα για τις επιχειρήσεις, το οποίο σημαίνει ότι έχουν μόνο μία εποπτική αρχή απέναντί τους επιχειρήσεις αντί για 28 και το ίδιο ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως της έδρας τους ή της σύστασή τους. Και οι επιχειρήσεις που βασίζονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εφαρμόζουν το ίδιο αυτό ρυθμιστική πλαίσιο και αυτό οδηγεί σε πιο ενοποιημένους και ισότιμους κανόνες. Για την τεχνολογική ουδετερότητα την την... το δικαίωμα μεταφοράς των δεδομένων από έναν πάροχο στο άλλον και αυτό σημαντικό, όπως και για τις μικρές και νέες επιχειρήσεις θα έχουμε λύσεις πιο φιλικές προς την προστασία της ιδιωτικότητας. Θα υπάρχει αυτό που ονομάζουμε ε, προστασία δεδομένων βάσει σχεδιασμό και ως βασική θέση που σημαίνει ότι ε, η τεχνολογία θα προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα από το σχεδιασμό της και ε, ως εξυποθέσεως. Επίσης η ανωνυμοποίηση και η κρυπτογράφηση έχουν συμπεριληφθεί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων Άλλη μια μάχη που εδώσαμε και νομίζω ότι καταφέραμε να κερδίσουμε στο τέλος ήταν για την επιστημονική έρευνα και την ιστορική έρευνα. Αρχικά είχαμε δύο περιορισμούς ε, στην ε, μεταχείριση των δεδομένων αλλά στο συμβαστικό κείμενο που αποκλείονται τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα από τις ε, περιορισμούς των διατάξεων του κανονισμού. Και αυτό συνολικά βελτιώνει την κατάσταση. Και τέλος, και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό για τις μικρές και μισές επιχειρήσεις που μας αφορά στην έτρε, αυτές θα επιφεληθούν από την ε, σημαντική μείωση των γραφειοκρατικών δικασιών. Είχαμε ένα κόστος για τις επιχειρήσεις άνω των 130 εκατομμυρίων ανά έτος σχετικά με τις πολλαπλές αρχές που έπρεπε να απευθύνονται. Δεύτερον, όταν η πρόσβαση δεδομένα είναι μη δικαιολογημένη και υπερβολική, θα επιβάλλονται κυρώσεις. Επίση, οι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει δεν θα έχουν υποχρέωση διενέργειας ε, αξιολόγηση αντικτύπου εκτό αν υπάρχει αποδεδειγμένο ψηλός κίνδυνο. Επομένως λοιπόν μετά από τρία χρόνια έχουμε πλέον τον κανονισμό μας και όταν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο όπως θα γίνει φαντάζομαι τον Απρίλιο θα είναι πλέον επίσημα νόμος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε κύριε Κέλλη για τη θαυμάσια αυτή δουλειά που κάνατε εξ ονόματος της Επιτροπής και επιτρέψτε να πω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η δουλειά. Μπορούμε να είμαστε όλοι περήφανοι για την προσωπική σας προσπάθεια όχι μόνο καλύψαμε την καθυστέρηση αλλά την ξεπεράσαμε. Η συνέχεια της συνάντησής μας είναι στις 3 ε, όπου θα έχουμε τη χαρά να δούμε τον Επίτροπο Μόερας αυτά προς το παρόν.